Σα Präsident. Vielen Dank. Σας ευχαριστώ. Ε, αρχίζει πάλι η συνεδρίαση. Παρακαλώ καθίστε. Τα πρακτικά είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγκρίνονται τα συνοπτικά πρακτικά. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα στην ημερή.